Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρία της Επιτροπής ε, Ρέτζι για σήμερα. Παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Ας έχουμε λοιπόν και λίγο ανοιξιάτικη διάθεση σήμερα. Ο ήλιος λάμπει έξω, ο καιρός είναι ωραίος, η άνοιξη έρχεται και η ζωή συνεχίζεται και δεν εξαρτάται από τις λεπτομέρειες που μας απασχολούν εμάς συνεχώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν να έχουμε μια παραγωγική και καλή συνεδρίαση σήμερα. Θα ξεκινήσω με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, σχόλια, συστάσεις, όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Κατόπιν, έγκριση των πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων συνεδρίαση από τις, για τις 14 Φεβρουαρίου και τις 20 Φεβρουαρίου του 2019. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο όπως γνωρίζετε. Προτείνω ως συνήθω, εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Τρίτο σημείο, ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω και πάρα πολλές ανακοινώσεις για σήμερα. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας στα αποτελέσματα της αποστολής μας στην Πορτογαλία που έγινε από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 1η Μαρτίου. Γνωρίζετε ότι ήταν η τελευταία αποστολή της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Επικεφαλής ήταν ο κύριος Βανίστερλο και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας πει δύο λόγια για τα αποτελέσματα της ε, αποστολής. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να σχολιάσουμε, διότι έχουμε, είχαμε μία πλήρη αποστολή, η εκπροσώπηση από τις διάφορες πολιτικές ομάδες δηλαδή, πλήρη συμμετοχή και στις επισκέψεις και από τα μέλη από την Πορτογαλία και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, διότι πολλές άλλες αντιπροσωπείες ε, δεν ε, έγιναν και μας ενδιαφέρουν λοιπόν ιδιαίτερα τα ε, αποτελέσματα αυτών που κάνουμε και η επίσκεψη αυτή στην περιοχή Νόρτε, στα βόρεια της Πορτογαλίας, δείχνουν ακριβώς τι κάνουμε και γιατί εργαζόμαστε. Αν έχεις μια περιφέρεια η οποία είναι σε πλήρη μετάβαση ε, πριν από 15-20 χρόνια ήταν επικεφαλής στην κλωστοϊφαντουργία, στα δέρματα και είχαν ε, εμπορικά σήματα γνωστά ε, και, εδώ και καιρό. Και λόγω του ανταγωνισμού χρειάστηκε να αναζητήσουν άλλες δραστηριότητες και άλλες πρωτοβουλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σήμερον ημέρα, ιδέως ε, ε και τις, για τις άλλες χώρες και τα μέλη που επισκέφτονταν από άλλες χώρες. Στην επίσκεψη είδαμε ότι αν υπάρχει ένα σταθερό και ε, ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο είναι αφαισιωμένο στις εφαρμοσμένες επιστήμες και σε ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να παράγουν προϊόντα, μπορούμε να έχουμε νέες πρωτοβουλίες οι οποίες είναι διαρκείας. Και διαπιστώσαμε σε αρκετούς τομείς, αλλά θα αναφέρω έναν, ε, νέες πρωτοβουλίες στην αυτοκινητοβιομηχανία, ε, οχήματα ε, χωρίς οδηγό και όλη η τεχνολογία που υφέρπει, ε, πολύ συχνά σκέφτεται κανείς στη Γερμανία. Αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνουν εκεί τα πράγματα και η αντιπροσωπεία μας είχε περιθώριο να... Ε, κάνει μια μικρή διαδρομή ε, σε αυτά τα ε, οχήματα. Είναι μια εταιρεία η οποία αποκαλείται Bosch, η οποία ε, με όλες τις πληροφορίες ασφαλείας. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε εκεί και από ενημέρωση από τις ε, περιφερειακές αρχές σχεδιασμού και από τους πολιτικούς ηθήνοντες, δημάρχους και δημοτικά συμβούλια αλλά επίσης και σε συζητήσεις μας με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπροσώπους ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, η περιφερειακή πολιτική είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη ε, τμήματων της χώρας θα υποβληθεί πλήρη έκθεση και μπορούν και οι συνάδελφοι να πούν την άποψή του. αλλά εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το γεγονό ότι μπορεί κανεί να ανακάμψει μέσω της ε, εφιούς εξειδίκευσης, γνωρίζοντας πού θα επενδύσουμε για 7-10 χρόνια και αυτό προσελκύει νέες δραστηριότητες. όπως είπα και στην αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, ε, στη γεωργία, την ποιότητα της πόλης του Πόρτο, την οποία επισκεφθήκαμε και είναι τουριστικός προορισμός, ε, πολιτιστική κληρονομιά επίσης και πολλά άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν εκεί. Ε, μου δόθηκε η αίσθηση προσωπικά ότι ήταν η καλύτερη ε, αντιπροσωπεία της οποίας θα μπορούσα να ηγηθώ, χάρη στα μέλη της και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η ενημέρωση λοιπόν για την αποστολή αυτή και θα ήθελα να πω ότι όλες οι ε, αποστολές που διοργανώθηκαν αυτή την πενταετία ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς και ιδιαίτερα χρήσιμες για το έργο της ε, Επιτροπής μας. Είχαμε διάφορα παραδείγματα από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα διάφορα <coughs> κράτη-μέλη, ε, διάφορα θέματα, διαφορετικές επιτυχίες, αλλά όλα αυτά οδήγησαν σε χρήσιμες γνώσεις ε, και ε, να διαμορφώσει άποψη η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Ευχαριστώ λοιπόν όλα τα μέλη που συμμετείχαν στις αντιπροσωπείες. Ένα πολύ σημαντικό σκέλος λοιπόν των εργασιών μας που ολοκληρώθηκε πλέον. Συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τον κανονισμό των κοινών ε, προμηθειών το CPR. Εγκρίθηκε η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια με κάποιες αλλαγές στις 13 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια ο φάκελος αναπέμφθηκε και πάλι στην Επιτροπή για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Έγιναν τρεις ε, συναντήσεις ε, στις 19 Φεβρουαρίου, στις 26 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου καθώς επίσης και μία σειρά από τεχνικές συνεδριάσεις σε επίπεδο προσωπικού. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρέλ αν θέλει να μας πει λίγο την εικόνα που έχει αποκομίσει για αυτούς τους τριμερείς διαλόγους και το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κυρία Κρέλη, έχετε το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι συμμετέχοντες στον τριμερή διάλογο ήθελα να ολοκληρώσουν ε, το σκέλος του προγραμματισμού. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να γίνουν τουλάχιστον οι τεχνικές συναντήσεις και ο τριμερής διάλογος. Στον τρίτο τριμερή διάλογο, το Κοινοβούλιο έφτασε σε ένα συμβιβασμό για, την, ε, το σύνολο της ε, δέσμης μέτρων, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο για μας. Συμβιβαστήκαμε, δώσαμε πράγματα, και πιστεύαμε πραγματικά πως το Συμβούλιο θα δεχόταν το συμβασμό αυτό. Μετά, αν κατάλαβα καλά, πήγαν τις ομάδες εργασίας τους, το συζήτησαν και γύρισαν λέγοντας ότι θέλουν και άλλο χρόνο. Δυστυχώ, νομίζω πω ε, πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι έχουν πάρα πολύ χρόνο μέχρι την έναρξη τη νέα περίοδου. Ε, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη αλήθεια αυτό. Και είναι πραγματικά κρίμα γιατί προσπαθήσαμε ε, όσο μπορούσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στήριξε ε, για να βρούμε αυτόν τον ε, συμβιβασμό. Η Προεδρία ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα αυτό, προσπάθησε και μετά τα κράτη-μέλη σταμάτησαν τη διαδικασία και τώρα είμαστε εκεί που ξέρετε. Θα ψηφίσουμε για την ολοκλήρωση του θέματος σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς συζήτηση, χωρίς τροπολογίες και μετά το επόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό στη συνέχεια. Ελπίζω λοιπόν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό θα γίνει από το νέο Κοινοβούλιο, από τη νέα Επιτροπή, με όποια μέλη και αν έχει. Η Επιτροπή μας ήταν η Προεδρεύουσα Επιτροπή στις ε, συζητήσεις, οπότε θα δούμε αργότερα μετά το καλοκαίρι τι θα γίνει αν τα κράτη-μέλη θα συνειδητοποιήσουν ότι ο χρόνος δεν είναι τόσο πολύ όσο νόμιζαν. Φαίνεται πως είναι πολύ. Όμως να πω ε, πως αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία που θα έχω για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή, τους ε, σκιώδεις εισηγητές να ευχαριστήσω όλους τους ε, πολιτικούς συμβούλους, τη γραμματεία, τους βοηθούς μας, διότι είχαμε πάρα πολλή δουλειά και εργαστήκαμε πολύ σκληρά για τις ε, νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Νομίζω λοιπόν πως κάναμε καλή δουλειά και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως ε, κομμάτι της προεκλογικής μας εκστρατείας, διότι η πολιτική συνοχή είναι το πρώτο που βλέπει ο πολίτης. Είναι το πιο ορατό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής στη δική τους ε, περιφέρεια, τη δική τους κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά και ελπίζω να δω αρκετούς από εσά και στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανίστελ έχει το λόγο. Ναι, είναι σωστά όσα είπες, όμως ε, θα σε ενημερώσω πως δεν θα επιστρέψω μετά τις ευρωεκλογέ. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε τη γνωμοδότησή μας εγκαίρως, έτοιμη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν και όσους συνεργάστηκαν γι' αυτό, όμως το Συμβούλιο δεν ήταν έτοιμο. Και είναι παράλογο να ακούμε από την ε, Ρουμανική Προεδρία να λέει πως πρώτη προτεραιότητά μας είναι η πολιτική συνοχή και μετά να ασχολούνται με τον ορίζοντα Ευρώπη, να έχουν συμφωνία. Μάλλον το ίδιο θα γίνει και με το Invest EU. Με όλα λοιπόν, εκτός από την πρώτη τους προτεραιότητα. Διαβάστε τις. Κυρία Κρέλη, λοιπόν, νομίζω πως ε, είστε ιδιαίτερα ε, ευγενική και προσεκτική με τις εκφράσεις σας. Εγώ δεν θα έλεγα το ίδιο, δεν συμφωνώ ε, με αυτά που άκουσα. Γιατί μην ξεχνάμε πως μας πίεσαν πάρα πολύ. Το Συμβούλιο είχε αρκετά προορατική στάση και βέβαια μετά τις ευρωεκλογές θα ξαναπιάσουμε το θέμα αυτό. Θα γίνει στην πρώτη ολομέλεια η συζήτηση για το θέμα σε πρώτη ανάγνωση. Και σίγουρα ελπίζω πως ε, θα συνεργαστούμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου μαζί μας. Θα θέλατε να σχολιάσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λοιπόν ευχαριστώντας και εγώ το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα εσάς κυρία Πρόεδρε και τους δύο συνεισηγητές για τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και πράγματι θεωρώ πως η κυρία Κρέλ συνόψισε πολύ καλά την όλη διαδικασία. Είχαμε ελάχιστο χρόνο, τρεις εβδομάδες. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το χρόνο όσο καλύτερα μπορούσαμε. Η Προεδρία κινητοποιήθηκε, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να σημειωθεί πρόοδος. Όπως όμως, ε, γνωρίζετε, στο Συμβούλιο έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε περίπου στα μισά μέχρι να υιοθετήσουμε την ε, γνωμοδότησή μας για τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Όπως ξέρετε υπάρχουν μπλοκ και μετά από δυόμισι μήνες έχει σημειωθεί πρόοδος για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να λάβουμε μία εντολή Και ίσω αυτός ήταν ο λόγος που δεν υπήρχε αρκετή ευελιξία από πλευρά κρατών μελών έτσι ώστε να δεχτούν κάποιες τροπολογίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να δούμε αποτελέσματα για τη συνοχή και έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Όπω ακούσατε και στην σχετική παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, στόχο των διαπραγματεύσεων είναι μια γενικότερη προσέγγιση όταν φτάσουμε στο τέλος των έξι μηνών. Θέλουμε λοιπόν πλήρη διαπραγματευτική εντολή, όχι μόνο για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, αλλά και για τα άλλα προγράμματα, το ESF+, το Interreg, μεταξύ άλλων. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αποτελέσματα και σχετικά με τους ε, τριμερείς διαλόγους να πούμε πως ε, η Ρουμανική Προεδρία έχει δουλέψει αρκετά ώστε δεν απέχουμε πολύ από την επίτευξη συμφωνίας και θα είναι πολύ εύκολο η επόμενη Προεδρία να φέρει πέρα σε αυτό που έχει ξεκινήσει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη στην προεκλογική σας εκστρατεία. Ευχαριστώ. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα, αλλά να αναφερθούμε και σε μία λεπτομέρεια ακόμα. Είναι σχεδόν η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής μας και θα είμαι ειλικρινής. Θα πω ότι αυτός ο αγώνας για την πολιτική συνοχή, αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται το φθινόπωρο. Διότι ο λόγος που δεν είχε σημειωθεί πρόοδος μέχρι τώρα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να δεχτούν τη συνολική εικόνα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. και τον πολύ σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής, τον οποίο καταφέραμε να διατηρήσουμε. Γι' αυτό νομίζω πως η Επιτροπή μας έκανε πολύ καλή δουλειά. Ετοιμάσαμε την έκθεση, την ψηφίσαμε για να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, όμως θα συνεχιστούν οι εργασίες στο φθινόπωρο. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι καλή επιτυχία στην επόμενη Επιτροπή Περιφυριακή Ανάπτυξης στις διαπραγματεύσει. διότι αυτό είναι ο λόγος της καθυστέρησης, η μη ετοιμότητα των κρατών μελών να δεχτούν όλα τα συστατικά στοιχεία της ε, πολιτικής συνοχή. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ θα ψηφίσουμε στη, τη συμφωνία περί διατάξεων σε πρώτη ανάγνωση την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα ψηφίσουμε επίσης και για άλλα ταμεία, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ίντερεγ, την επόμενη εβδομάδα επίσης στο Στρασβούργο, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας για τα θέματα τα οποία έχουμε αναλάβει. Αυτά λοιπόν προς ενημέρωσή σας για το θέμα αυτό και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Μόνο μία ψηφοφορία έχουμε, η τελευταία έχει να κάνει με την προσαρμογή της προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 με 2023. Ο κύριος Πιοτρόφσκι είναι εισηγητής. Εμείς είμαστε η αρμόδια επιτροπή. Δεν έχουμε λάβει γνωμοδοτήσεις από τις συνδεδεμένε επιτροπές, ε, προπολογισμού, απασχόληση και αλληλεία. Αποφάσισα να μην καρταρτήσουν η γνωμοδότηση. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να εγκρίνουμε, να ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο έκθεσης. Κύριε Πιετρόφσκι, θέλετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Την προηγούμενη φορά έγινε ανταλλαγή απόψεων και διαβουλευτήκαμε όχι μόνο με τα μέλη της Επιτροπής μας, αλλά και με εκπροσώπους των κρατών μελών. Το επίπεδο ήταν στο 3% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε το 1% και στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μετά τις διαβουλεύσεις κατέληξε στο 2%. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξουμε το ποσοστό αυτό και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεδεθειμένη να αποδεχτεί το επίπεδο αυτό του 2%. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιετρόφσκι, λέει πρόεδρος. Έχετε το κατάλογο ψηφοφορίας μπροστά σας. Είναι και σύντομο άλλωστε. Περίεργο αυτό για μας. Και τώρα να περάσουμε κατευθείαν στις τροπολογίες 2 και 3 οι οποίες είναι και ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εδώ θα χρειαστεί νο, ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε μια και πρόκειται για ψηφοφορία κλειδί. Για την τροπολογία 1 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ, έλεγχος. Πέρα. Εγκρίνεται. Και τώρα να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση με πλήρη ε, πλειοψηφία, με όλες τις ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στον κύριο Πιτρόφσκι. Uh, στην Ολομέλεια θα ψηφίζουμε στην πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου. Θα περάσει στην Ολομέλεια λοιπόν η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Did you take your time? Yes, thank you. Thank you. We continue Να συνεχίσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης για τους κανονισμούς, ε, εφαρμοστικός κανονισμός ε, για την 13.03 του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη μορφή της χρηματοδότησης που δεν σχετίζεται με το κόστος των σχετικών ε, επιχειρήσεων. Τεχνικό το θέμα Αυτή η πράξη καταξιοδότηση ε, μα συμπληρώνει τον κανονισμό και λαμβάνει υπόψη τις αλλαγέ που έγιναν στο CPR για το 2014-2020 από τον κανονισμό Omnibus. Αποτελεί ουσιαστικά μια συνέχιση των ε, αποφάσεών μας στο Omnibus. Η προθεσμία για ενστάσεις σε ό,τι αφορά το ψήφισμα της Ολομέλειας είναι η 15η Απριλίου ενδεχόμενη παράταση για τα δύο μήνε. Η συνήθιστη διαδικασία δηλαδή. Και τώρα θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα παρουσιάσει το σχέδιο πράξη κατά να δώσω το λόγο στους συντονιστές και στα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια, αν θέλουν να σχολιάσουν ή να κάνουν ερωτήσεις και στην... στο τέλος θέλουμε να λάβουμε και την απόφαση για την ε, απόφαση αυτή, για την πράξη καταξιοδότηση. Η κυρία Βάγνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής. Να, καλωσορίσω και, να καλημερίσω και την Πρόεδρο. Να σας ευχαριστήσω που μας αφαιρώνετε το χρόνο για να εξετάσουμε το θέμα αυτό, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ τεχνικό. Δεν θα σας κουράσουμε με λεπτομέρειες όμως. Να υπενθυμίσω μόνο το ιστορικό του φακέλου Omnibus αυτή η πράξη κατά εξουσιοδότηση ουσιαστικά εντάσσεται στην όλη ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στα μέσα Σεπτεμβρίου 2016 με σκοπό να δώσει απάντηση στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και των δικαιούχων και των κρατών μελών που ζητούσαν ε, επιγόντως απλοποίηση. Αυτή η πρωτοβουλία, λοιπόν, η Omnibus, ήταν μια στοχευμένη πρωτοβουλία η οποία έγινε με σκόπο να μην ανατραπούν οι υφιστάμενοι κανόνες και να υπάρξει πρόβλημα στην ε, υλοποίηση, η οποία πήγαινε αρκετά ομαλά. Θέλαμε απλά να απλοποιήσουμε κάποια στοιχεία. Αυτή λοιπόν η πράξη κατά εξουσιοδότηση έχει ως σκοπό να δώσει μία νέα μορφή, αν θέλετε, επιδοτήσεων, ενισχύσεων που να μην σχετίζεται με το πραγματικό κόστος. Και αυτό γιατί χρειάστηκε. Γιατί ήταν σημαντικό. Γιατί ένα από τα νέα στοιχεία της ε, πρότασης Omnibus ήταν να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται πληρωμές που να μην σχετίζονται με το κόστος αλλά για να χρηματοδοτηθούν κάποιες συνθήκες. Άρα, το θέμα ήταν να γίνει η πληρωμή αυτή όταν συντρέχαν οι προϋποθέσεις αυτές, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να τηρούνται πρακτικά και λογαριασμοί για το κόστος, το πραγματικό της κάθε επιχείρησης. Γιατί είναι σημαντικό λοιπόν αυτό, είναι τεχνικό στοιχείο, αλλά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία αποτελεί μια μεγάλη απλούστευση, γιατί επικεντρωνόμαστε στο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να πετύχει κάθε επιχείρηση. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν υπήρχαν και συντρέχαν οι προϋποθέσεις επί των οποίων είχαμε συμφωνήσει με τα κρατη όσο και να είχαν κοστίσει, μπορούσαμε να ζητήσουμε, να ζητηθεί δηλαδή επιστροφή, αποζημίωση. Και έτσι λοιπόν απλοποιείται ο συνολικός μηχανισμός. Η πρωτοβουλία αυτή έπρεπε να μετατραπεί και σε νομοθετική πράξη, αυτή την πράξη κατά εξουσιοδότηση, η οποία είναι πολύ σύντομη, μόνο τέσσερα άρθρα. Έχει ένα παράρτημα λίγο πιο λεπτομερές και ουσιαστικά εξηγεί με λεπτομέρεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ισχύσει το σύστημα αυτό. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής οι τομεί στου οποίου ισχύει η πράξη καταξιοδότηση είναι μέτρα, είναι μέτρα για την ενεργειακή αποφατικότητα και για την ενεργειακή απόδοση. Περιλαμβάνει και όρους για το πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση και περιλαμβάνεται και περιγραφή του κανόνων για τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις που θα πρέπει να γίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ότι ο έλεγχος θα γίνεται αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τις συνθήκες χρηματοδότησης, τους όρους χρηματοδότησης. Αυτό θα ελέγχεται και μετά θα γίνεται η αποζημίωση. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη περίπτωση που έχει να κάνει με το ERDF και το Ταμείο Συνοχής, στην προκειμένη περίπτωση. Και νομίζω ότι με τα στοιχεία αυτά κάλυψα τα βασικά στοιχεία και τους βασικούς νεοτερισμούς σε ό,τι αφορά την πρότασή μας. Θα βάλω τελεία λοιπόν εδώ και δεν θα μπω σε υπερβολικές τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες έτσι και αλλιώς θα πρέπει να ελέγξουν οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη για να κατανοήσουν και να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. Να σας αναφέρω απλά ότι την πρόταση αυτή την παρουσιάσαμε στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου προ Έγινε μια διαβούλευση με του συμπρεγνώμονε των κρατών μελών τον προηγούμενο Νοέμβριο. Και στις 15 Φεβρουαρίου 2019 εγκρίθηκε ο φάκελο αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και για τον χρόνο σα. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Πολύ σαφής η εξηγήση σας. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο τώρα. Έχετε κάποια ερώτηση, έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Κάποια ένσταση να εκφράσετε. Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχει λοιπόν οποιαδήποτε αντίρρηση, όλα είναι σαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξηγήσεις αυτές. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, για την πράξη αυτή κατά εξουσιοδότηση. Ολοκληρώθηκε η εξέταση του θέματος. Δεν θα χρειαστούμε λοιπόν τους δύο μήνες για υποβολή ενστάσεων. Θεωρείται ολοκληρωμένο το θέμα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λέο Μπρίνκατ, μέλος του Εκτικού Συνεδρίου. You know that we Ξέρετε ότι έχουμε πολύ επικοδομητική συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουν γίνει πολλές ανταλλαγές απόψεων, λάβαμε πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες από τα μέλη του δικαστηρίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους για την καλή συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με χαρά σήμερα καλωσορίζω τον κύριο Μπρινκάτ, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα παρουσιάσει την ειδική έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ξέρετε ότι έγιναν πολλές συζητήσεις για το Ταμείο αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και τις ε, θέσαμε και στους εκπροσώπους ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και τώρα ε, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσουμε και τα πορίσματα της έκθεσής σας. Θα δώσω πρώτα το λόγο σε εσά για ένα τέταρτο 20 λεπτά να μας παρουσιάσετε την έκθεση, αλλά πρέπει να αναφέρω ότι εδώ στην συνεδρίαση έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Ίσως ε, να είναι καθοδόν. Διότι σκοπεύαμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλουμε να ακούσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Να ξεκινήσουμε όμως με την παρουσίαση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχετε το λόγο, κύριε Μπρινκάτ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κυρία Μιχαέλοβα, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά να σας ε, παρουσιάσω σήμερα την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ε, τις δράσεις που χρειάζεται για να επιτύχει πλήρως. Αυτός ήταν ο πλήρης τίτλος της έκθεσης, ε, μαζί φυσικά με τις απαντήσεις της Επιτροπής παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος μας δεν τονίζει τις ιδιαιτερότητες σε περιφερειακό επίπεδο των δράσεων του Ταμείου, κάποια από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται, τα οποία αφορούν και τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν και το ρόλο των ε, ε, τοπικών τραπεζών, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και εθνικών τραπεζών, είναι πολύ σημαντικές σε περιφερειακό επίπεδο. Το ΕΦΣΙ συστήθηκε το 2015 ως τμήμα του Σχεδίου Επενδύσεων για την Ευρώπη και σχεδιάθηκε για να αντιμετωπίσει το κενό επενδύσεων που προέκυψε από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Όπως γνωρίζετε καλά συνέβη το 2008 και έπληξε πολύ ε, σκληρά τις περιοχές ε, και τις περιφέρειες ε, της Ευρώπης. Ε, συστήθηκε εντό τη Τράπεζα Επενδύσεων και ξέρετε ότι υπήρχε μια διευθύνουσα επιτροπή και ε, συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, δόθηκαν 16 ε, δι εγγύηση στον προπολογισμό και 5 δι από τις ίδιου πόρου τη Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο να κινητοποιήσουμε επιπλέον 315 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση μέχρι τον Ιούλιο του 2018 στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτουν τομείς πολιτικής και όλα τα κράτη-μέλη. Ο στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογήσουμε κατά πόσον το Ταμείο ήταν αποτελεσματικό, κατάφερε να ε, συλλέξει πόρους για να υποστηρίξουν επιπλέον επενδύσεων, επενδύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύφθηκαν οι επιχειρήσεις από την έναρξη του Ταμείου το 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Ω τμήμα του ελέγχου μα, είδαμε εκθέσεις για, την, ε, για τις επιδόσεις του Ταμείου που δημοσιεύθηκαν μέχρι να γίνει ο ελεγχός μας. Εξετάσαμε το χαρτοφυλάκιο επιχειρήσεων του ΕΦΣΥ, είδαμε και ε, κάποια δείγματα επιχειρήσεων και υπήρξαν και συνεντεύξεις ε, και επαγγελματιών από το, το Ταμείο και από την Τράπεζα Επενδύσεων. Και επιπλέον διαβουλευτήκαμε και με πολλούς ενδιαφερομένους τον Ombudsman για να έχουμε μια εικόνα για την προσέγγιση, την Επιτροπή των Περιφερειών και επίσης και την ΕΟΚΕ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Κάποια στιγμή συναντήθηκα και προσωπικά με αρκετούς ευρωβουλευτές ε, και που ενδιαφέρθηκαν για το Ταμείο Στρατηγικής Ανάπτυξης ε, για να ξέρουμε και τη δική τους την οπτική για το θέμα. Και ευχαριστώ πολύ όλους εκείνους που συναντήσαμε γι' αυτό διαπιστώσαμε ότι είχαμε καταφέρει να έχουμε έγκριση πάνω από 59 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συγγνώμη, επενδύσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2018 ε, και επιπλέον είχαμε 65,5 δις ε, μέχρι τις 17 Ιουλίου του 2018. Πολλοί παραγόντες συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα ε, κυρίως το γεγονός ότι υπήρχε η εγγύηση προπολογισμού που δίνεται στην ε, Τράπεζα Επενδύσεων, υπήρχε ευελιξία, υπήρχαν ελάχιστοι στόχοι και περιορισμοί για το χαρτοφυλάκιο του ΕΦΣΥ, ε, υπήρχε ε, μια οργανωμένη ε, διακυβέρνηση και συνεργασία με εθνικές τράπεζες και ιδρύματα. Η στήριξη του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μας βοήθησε να επιτευχθούν στόχοι και να ε, ε κάνουμε ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλότερου κινδύνου για το ΕΦΣΥ. Ωστόσο, κάποιες ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που υπεγράφησαν από το, η Τράπεζα Επενδύσεων ήταν χαμηλότερες από όσο προβλεπόταν. Υπήρχαν και κλασικά παραδοσιακά δάνεια που προσφέρονταν και ε, ήταν εξασφαλισμένοι όλοι οι δανειστές ε, και υπήρχαν και εταίροι υψηλότερου κινδύνου και είδαμε και τι ακριβώς μπορούσαν να γίνουν για άλλα διαθέσιμα υψηλού κινδύνου χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης, εν μέρη, ε, αντικαταστάθηκε χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαχειριζόμαστε κεντρικά ε, στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Η ανάγκη λοιπόν που υπάρχει είναι η Επιτροπή και η Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσουν πιθανές επικαλύψεις μεταξύ των επιχειρήσεων και τη, ο παράθυρο της καινοτομίας και τα ευρωπαϊκά ε, διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Να πω ότι δεν υπάρχουν προφανείς επικαλύψεις μεταξύ του ΕΦΣΥ και τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάσαμε. Ε, ξεκινήσανε μεγαλύτερα έργα υποδομών μέσω του ΕΦΣΥ που συνήθως δεν καλύπτονται από αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Εκεί έχουμε πιο περιφερειακά και μικρότερα έργα. Ε, επειδή όμως θα υπάρξουν ε, πιέσεις προς το τέλος της χρηματοπιστωτικής περίοδου, μπορεί να στοχεύσουμε και σε αυτές τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Το γεγονός ότι ε, θεωρήθηκαν ότι οι διαδικασίες του ΕΦΣΙ προσφέρουν κάποια πρόσθετα στοιχεία ε, και θεωρούμε ότι έχουμε κάποια στοιχεία υψηλού κινδύνου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση από άλλες πηγές για ένα έργο. Τα αποτελέσματά μας είναι ότι το 1 τρίτο των υποδομών ε, και των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το Innovation Window θα μπορούσαν να είχαν γίνει και χωρίς τη στήριξη του ΕΦΣΥ η επιλογή του ΕΦΣΙ ήταν είτε γιατί ήταν ευθυνότερο είτε γιατί παρήχε και μεγαλύτερες εγγύησεις. Διαπιστώσαμε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες κάποια έργα θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικούς φορείς ή από την Τράπεζα Επενδύσεων στις συνήθεις διαδικασίες με τα συνήθη κονδύλια. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμήσουμε το, ε, την επένδυση που κινητοποιήθηκε ε, ορισμένες φορές ήταν υπερβολική ε, και ο παράγοντας πολλαπλασιασμού ορισμένες φορές περιλαμβάνεται και εκφράζει κάτι ως πολλαπλάσιο ε, της επένδυσης που έγινε. Ε, οι εκθέσεις ε, της Τράπεζας Επενδύσεων περιλαμβάνουν όλες τις επιλέξιμες επενδύσεις που έγιναν, ανεξάρτητα από το μερίδιο το οποίο κινητοποιήθηκε από το ΕΦΣΥ. Και αυτό το φαινόμενο της πολλαπλασιαστικής ε, ε επένδυσης ε, διαπιστώσαμε ότι μάλλον δηλώνεται σε υπερβολικό βαθμό. Επίσης ε, υπάρχει κίνδυνος ακριβώς ε, επειδή έχουμε διαφορετική χρηματοδότηση να έχουμε διπλή καταμόρτιση όταν, ε, καταμέτρηση συγγνώμη, όταν υπολογίζουμε την επένδυση και τον πολλαπλασιαστικό παράδειγμα. Το γεγονό ότι δεν έχουμε συγκρίσιμη επίδοση και οι δείκτε για την παρακολούθηση και τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις εγγυήσεις στον προπολογισμό μειώνει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Ε, το χαρτοφυλάκιο του ΕΦΣΙ στο τέλος του 2017 ήταν εντός των ενδεικτικών ωραίων που είχαν καθοριστεί για την επένδυση σε συγκεκριμένους τομείς. Αλλά η γεωγραφική συγκέντρωση του ΕΦΣΙ και οι επιχειρήσει οι οποίε υπεγράφησαν δεν ήταν επαρκώς ισορροπημένοι και συνήθως κατέληξε ε, σε κάποιες από τις μεγαλύτερε 15 χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι χώρες οι οποίες πήραν τις μεγαλύτερες επενδύσεις ήταν αυτές οι οποίες είχαν τις πιο ανεπτυγμένες εθνικές τράπεζες και ιδρύματα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη και τεχνική συνδρομή σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι τόσο ανεπτυγμένοι. Αυτό το διαπιστώνουμε με λεπτομέρεια στα στοιχεία της έκθεσης, ε, στη σελίδα 87 και στην παράγραφο 84 της έκθεσης. Κατά την άποψή μας, εάν ε, οι συμβουλευτικοί κόμβοι είχαν υποστηρίξει λίγο καλύτερα και είχαν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα ε, τις δυνατότητες πόρων και χρηματοδότησης, θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα ευθύς εξ αρχής. Επιπλέον, επειδή δεν λάβαμε πληροφορίες για το πόσα ε, προγράμματα περίφθησαν, δεν μπορούμε να σας πούμε πώς ακριβώς έχει η γενικότερη εικόνα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ΕΦΣΙ ήταν αποτελεσματικό στη συγκέντρωση κονδυλίων για να έχουμε επιπλέον επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ουσιαστικές. Αλλά η εκτίμηση των επενδύσεων που κινητοποιήθηκε δεν λαμβάνει υπόψη και το γεγονό ότι κάποιε από τι επιχειρήσει του ΕΦΣΥ αντικατέστησαν άλλε επιχειρήσει τη Τράπεζα Επενδύσεων και ε, χρηματοπιστωτικά μέσα τη Ένωση ή το γεγονός ότι η στήριξη της ΕΦΣΥ πήγε σε προγράμματα τα οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές, ε, σίγουρα βέβαια με διαφορετικούς όρους. Επιπλέον πρέπει να λάβουμε μέτρα για να βελτιώσουμε τη γεωγραφική εξάπλωση του ΕΦΣΥ ε, και τις επενδύσεις που υποστηρίζει και να παρέχεται τεχνική συνδρομή στις εθνικές αρχές ε, και στις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές και σε περιφερειακό επίπεδο και το είδαμε αυτό και στις επαφές που είχαμε με διαφόρους ευρωβουλευτές. Καλούμε λοιπόν για μεγαλύτερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την προσβασιμότητα, να ενισχύσουμε το επίπεδο των πληροφοριών, να υπάρχουν στοχευμένες πληροφορίες για τις περιφερειακές αρχές ε, και εκπαίδευση για αυτούς που δεν έχουν αρκετή εμπειρογνωμοσύνη και στήριξη για την κατάρτιση των φακέλων προς υποβολή. Και το λέω αυτό όχι μόνο γιατί αναφέρομαι σε μια, απευθύνομαι συγγνώμη, σε μια Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι σημαντικά τα περιφερειακά θέματα ε, γιατί είναι πολύ περίπλοκη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΦΣΥ. Θα προτείνουμε λοιπόν να προωθήσουμε την ε, ε, αιτιολογημένη χρήση των προϊόντων της ε, Τράπεζας Επενδύσεων Υψηλότερου Κινδύνου υπό το ΕΦΣΥ, να ενθαρρύνουμε τη συμπληρωματικότητα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις εγγύησεις στον προπολογισμό. Τρίτον, να βελτιώσουμε την αξιολόγηση για το κατά πόσον κάποια έργα θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές. Τέταρτον, να εκτιμήσουμε καλύτερα την επένδυση που κινητοποιήθηκε και να βελτιώσουμε τη γεωγραφική εξάπλωση των επενδύσεων που υποστηρίστηκαν από το ΕΦΣΥ. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα Επενδύσεων. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι η Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκαν και τις πέντε συστάσεις μας ε, και σύμφωνα με αυτούς και πάλι, δύο από αυτές έχουν ήδη εφαρμοστεί. Υποθέτω το δεύτερο και το τρίτο. Η συνεδρίαση αυτή έχει μεγάλη αξία για τα θέματα που μας αποσχολούν και γιατί αυτό. Διότι επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στους συναδέλφους και στους εταίρους που συναντήσαμε, ότι όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η δημοσίευση της έκθεσης ναι μεν είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδικασίας, είναι αρχή της διαδικασίας. Θα παρακολουθούμε ε, στη συνέχεια πώς εφαρμόζονται οι συστάσεις μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους, ε, στα μέλη μας, αλλά πιο πριν ε, στον κύριο Ελπίν, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπρινκά, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε στην ΕΤΕΠ τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτήν την συνεδρίαση με θέμα το, την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνέδριου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας το, την ελεκτική ομάδα, αλλά και ε, τα μέλη της Επιτροπής για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε πριν τη δημοσίευση της έκθεσης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων οδεύει προς το στόχο κινητοποίησης τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία μέχρι το 2020. Ο στόχος ε, για τα 350 εκατομμύρια μέχρι το 2018 εκπληρώθηκε και με το παραπάνω. Σήμερα το ε, ποσό επενδύσεων έρχεται στα 390 εκατομμύρια ευρώ και η προσθετικότητα βρίσκεται στο κέντρο αυτή τη επιτυχία. Διότι έχουμε δει πω ε, δεν θα μπορούσε η ΕΤΕΠ να χρηματοδοτήσει τα project αυτά χωρί την δυνατότητα ε, που, τις δυνατότητες που έδινε το ΕΦΣΥ. Το Ταμείο λοιπόν αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΕΠ να αυξήσει τις επενδύσεις σε ε, προγράμματα υψηλού κινδύνου. Πριν το ΕΦΣΥ η ΕΤΕΠ μπορούσε να χρηματοδοτήσει ελάχιστες μόνο ε, επενδύσεις υψηλού κινδύνου, μόνο το 6% της συνολικής χρηματοδότησης δηλαδή που έδινε. Και χάρη στο Ταμείο αυτό τώρα το 30% των επενδύσεων μπορεί να ταξινομηθεί κάτω από τις ειδικέ δραστηριότητες. Το 75% περίπου των πελατών της ΕΤΕΠ είναι νέοι εταίροι της. Και τέλος, το 25% των ε, προγραμμάτων του ε, ΕΦΣΙ συγχρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε τις ε, ίδιες αρχές λειτουργίας και να στηρίξουμε την συνέχεια της ε, πρώτης φάσης του ΕΦΣΕ, το 2015 δηλαδή στο 2018. Χρειάζεται να δοθεί παράταση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, να υπάρξει ένα δεύτερο τέτοιο ταμείο στα πλαίσια του επόμενου πολιτου δημοσιονομικού πλαισίου που θα ξεκινήσει μετά το 2020. Ο σχετικός κανονισμός ε, για το ΕΦΣΥ θα καλύψει τα αρχικά στάδια της μετάβασης. Μετά, οι περισσότερες ανησυχίες του ηλεκτρικού συνεδρίου βρίσκουν απαντήσεις στην πρόταση για το ΕΦΣΙ 2. Ορισμένες πτυχές μάλιστα ήδη έχουν εφαρμοστεί, όπως είπε και ο κύριος Μπρινκά. Για παράδειγμα, οι συστάσεις σχετικά με την βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου χρηματοδότησης προγραμμάτων αλλά και η μέθοδος πολλαπλών υπολογισμών. Εδώ έχουν ήδη σημειωθεί βελτιώσεις σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποφευθούν οι επικαλύψεις. Τον Οκτώβριο του 2018 άρχισε να χρησιμοποιείται η νέα ε, μεθοδολογία η οποία ε, πρώτο παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για το δεύτερο στάδιο του ΕΦΣΥ. καταγράφονται οι περισσότερες ε, χρηματοδοτικές ενέργειες σύμφωνα με τις αναθεωρημένες ε, λειτουργίες. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεχίσει να προσπαθεί για καλύτερη κατανομή των πόρων σε προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατευθύνει τη χρηματοδότηση εκεί που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Χρειάζεται όμως να δούμε και τις θετικές εξελίξεις. Είναι φυσικό και λογικό το μέγεθος μιας οικονομίας να καθορίζει το μέγεθος ε, των επενδύσεων που στηρίζει η ΕΤΕΠ. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπολογίζουμε μόνο τον όγκο των επενδύσεων όταν εξετάζουμε τη γεωγραφική κατανομή των, ε, της χρηματοδότησης. οι αρχικές επενδύσεις του ΕΦΣΙ σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν πάρα πολύ κοντά. Όμως τελευταία έχουν αυξηθεί κατά πολύ αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως οι επενδύσεις γίνονται ολόνα και περισσότερο στα μικρά ε, κράτη-μέλη και σε εκείνα που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η Ελλάδα και η Εστονία είναι οι χώρες που εκπροσωπούνται περισσότερο ως προς την ε, κινητοποίηση χρηματοδότησης. Η Βουλγαρία και η Ισπανία είναι οι επόμενες χώρες στις οποίες γίνονται πολλές επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν για πολύ καιρό προσπάθησε να ε, βελτιώσει την ε, ισορροπία της γεωγραφικής κατανομής χρηματοδότησης μέσω ε, των ε, επιτόπου συνεργατών έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες της κάθε χώρας. Επίσης, υιοθετήσαμε διάφορα μοντέλα ενισχυμένης συνεργασίας που μας επέτρεψαν ε, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Αυτό εν μέρη χάρη στην, στον συμβουλευτικό κόμβο που χρησιμοποίησαμε. Επίσης, να είστε σίγουροι πως η ΕΤΕΠ συνεχίζει την προσπάθεια να εντοπίσει ευκαιρίες χρηματοδότησης χρέους εκεί όπου υπάρχει λόγος. Αυτά λοιπόν από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι λοιπόν, ακούσαμε και τις δύο πλευρές και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσίαση και την καλή συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μόνο δύο συντονιστές παρόντες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο εκτό από του ε, συντονιστέ και σε όσου έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Τσέλερ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπρίνκατ. Ευχαριστώ πολύ και ε, όλους τους συναδέλφους από το Ελεκτικό Συνέδριο που περίμεναν αρκετό καιρό έτσι ώστε να ε, δημοσιευτεί αυτή η έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων το ελεκτικό συνέδριο είναι πάντα επιφυλακτικό και συντηρητικό στις εκθέσεις του, γι' αυτό βλέπουμε ότι πάντα είναι και πολύ ακριβές. Βλέπω όμως ότι αυτά τα μεγάλα σχέδια που ανακοινώθηκαν είχαν λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα. Προέρχομαι από μια περιοχή στην οποία έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα στραβά, πάρα πολλά έργα τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν, ξεφούσκωσαν, θα έλεγε κανείς. και βλέπουμε ότι χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ε, ευρώ έργα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τεράστια ε, ε, έργα offshore για φυσικό αέριο, για μεταφορά ενέργειας και βλέπουμε ότι πάρα πολλές τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να χρηματοδοτήσουν παρόμοια προγράμματα. Προγράμματα τα οποία δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου. Επίσης, έχουν ε, χρηματοδοτηθεί προγράμματα με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία νομίζω πως ε, μπορούμε να τα θεωρήσουμε τουλάχιστον περίεργα. Για παράδειγμα, χρηματοδοτήθηκε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούσε ζωμό κότας για ζωοτροφή στις αγελάδες. Και πολλά άλλα τέτοια αστεία πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν κατάφερε με τη βοήθεια του ΕΦΣΙ να αυξήσει τη χρηματοδότησή της όμως, ο σκοπός ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ήταν άλλος. Ήταν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που είχαν πραγματικό νόημα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ πως θα πρέπει να επιστρέψουμε στον αρχικό μας στόχο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κράλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Την έκθεση ακόμα δεν την έχω διαβάσει. άκουσα μόνο τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου, τον κύριο Μπρινκ. Και νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Τσέιλερ είναι σωστά. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα φίλο των επενδυτικών αυτών προγραμμάτων και τα αποτελέσματα τα οποία μα παρουσιάσατε δεν μπορώ να πω ότι με πείθουν για να αλλάξω γνώμη. Και να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι τα χρήματα αυτά βγήκαν από τον ορίζοντα, από την διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης. Δεν ξέρω ε, τα προγράμματα αυτά, υποτίθεται ότι θα τα ενισχύαμε. Πέρα από αυτά που κάναμε με το πρόγραμμα στρατηγικών επενδύσεων, το ΕΦΣΙ, και ακούγοντας όλα αυτά στη συνέχεια, τα αριθμητικά στοιχεία μου προκαλούν έκπληξη και μας λέτε ότι τα στατιστικά στοιχεία επιδέχονται ερμηνεών. Όλα αυτά είναι καλά και ωραία για χώρες στο επίπεδο 92% του ΑΕΠ να υπάρχουν τέτοια προγράμματα δηλαδή εκεί. Αλλά προφανώς και η γεωγραφική κατανομή δεν στέκει απόλυτα. Το μόνο λοιπόν που έχω να πω είναι το εξής. Ελπίζω, ελπίζω το FC και το InvestEU, το διάδοχο πρόγραμμα, να είναι λίγο πιο σωστό και λίγο πιο σκόπιμο από το FC. αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση, θεωρώ, με το CPR. Ουσιαστικά πρέπει να πω ότι επιβεβαιώθηκαν όλοι μου οι φόβοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλετιτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την εξαιρετική έκθεση. Όλα όσα μας παρουσιάσατε στην έκθεση συνάδουν και με τις συζητήσεις μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, γιατί εξ αρχής αναρωτιόμαστε και συζητούσαμε κατά πόσον θα χρηματοδοτούσαμε τέτοια προγράμματα, κατά πόσο το ΕΦΣΙ θα υποκαθιστούσε ουσιαστικά χρηματοδότηση των Ταμείων Συνοχής και σε τελική ανάλυση είδαμε και με την εφαρμογή του ΕΦΣΙ τι συνέβη. Άρα η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ε, με την δρομολόγηση των ε, προγραμμάτων. Γιατί θυμόμαστε ότι στην αρχή και η Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέλεγαν ε, διάφορε ιδέε για δρομολόγηση τελικά των ε, συγκεκριμένων προγραμμάτων. Στην τελική ανάλυση, τι χρηματοδοτήθηκε, χρηματοδοτήθηκαν επικίνδυνα προγράμματα όπου δεν μπορούσε να γίνει, υπάρξει με άλλο τρόπο χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό αυτό για να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσουμε με το ΕΦΣΥ ή όχι και κατά πόσον έχουμε σε τελική ανάλυση επαρκή προγράμματα. Εγώ θεωρώ ότι το ΕΦΣΥ χρειάζεται. Υπάρχει ένα χάσμα τεράστιο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Θα πρέπει να το καλύψουμε. Δεν αρκεί ούτε η συνοχή, ούτε τα υπόλοιπα προγράμματα και ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προπολογισμού της Ένωσης. Είναι καλό λοιπόν να υπάρχει αυτή η συμπληρωματικότητα με τις ιδιωτικές επενδύσεις και να υπάρχει και ο πολλαπλασιαστικός παράγοντα αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τα πιο επικίνδυνα προγράμματα και σε ό,τι αφορά τη δρομολόγηση των προγραμμάτων. Το άλλο θέμα τώρα είναι η γεωγραφική κατανομή. Γιατί το είπαμε αυτό και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΕΤΕΠ, ότι πάνω από το 50% των χρηματοδοτήσεων ουσιαστικά πάνε στα πέντε μεγάλα κρατημέλη. Όταν λοιπόν κάνουμε μια ανάλυση των συνολικών ε, δραστηριοτήτων και πάλι στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Στην ΕΤΕΠ λοιπόν δεν μπορείτε να μας λέτε ότι ναι, αλλά όταν βάζουμε και τα υπολογίζουμε βάση ΑΕΠ είναι διαφορετική η εικόνα που προκύπτει. Ναι, αλλά ο δικό σα ο ρόλος είναι σύμφωνα με τη συνθήκη να μειώσετε τις ανισότητες να τι εξαλείψετε μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορείτε να τα μαγειρεύετε για να παρουσιάσετε μια διαφορετική εικόνα για το πώς θα πάνονται οι πόροι. Θα πρέπει τελικά να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ε, αρκετές χρηματοδοτήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτές θα πρέπει να υποστηρίξετε ως ΕΤΕΠ και να υπάρχει σωστή γεωγραφική ισορροπία σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φανίστελ Ροϊ. Έχει τώρα το λόγο, λέει ο πρόεδρο, Ναι, να προσθέσω και εγώ σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Το πήρα στα χέρια μου κατευθείαν όταν μας το υποβάλλατε πριν από ένα μήνα, νομίζω. Και πολλά από τα σημεία τα οποία είχαμε αναφέρει στο παρελθόν τα ξαναβρήκα. Αναγνώρισα τον τρόπο λειτουργίας σας. Πρώτη παρατήρηση. Γιατί έρχεται τώρα αυτή η έκθεση. Μόλις τελειώσαμε την πρώτη ανάγνωση και τη διαπραγμάτευση για το EU Invest πολλά αναγνώρισα από τα στοιχεία τα οποία ήδη λάβαμε υπόψη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά αναρωτιέμαι. γεωγραφική κατανομή, για παράδειγμα, και ισορροπία. Ποτέ αυτό δεν ήταν στους στόχους μας, αλλά το κάνουμε. Πλέον. Αν λοιπόν τέτοια επιρροή ασκείται, ε, θα συγχαίρω. Κατά δεύτερον, γιατί τη συμπληρωματικότητα μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη το γεγονό ότι άκουσα κάποιον να λέει ότι πρόκειται για χρηματοδότηση συμπληρωματική προ την Τράπεζα Επενδύσεων. Πολύ ωραία, αλλά δεν ήταν αυτή η συμπληρωματικότητα που είχαμε κατά νου. Το θέμα ήταν οι οικονομίε, οι επιχειρήσει που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά. Μα μιλάμε για συμπληρωματικότητα ή κινητικότητα τελικά. Τελευταία παρατηρήση. Είχα την αίσθηση ότι η έκθεση σας πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά κατηγορείται ότι βάζει επιπρόσθετα στοιχεία εδώ και εκεί, ε, δίνει χρήματα στην οικονομία και δεν υπάρχει ουσιαστικά σχέση μεταξύ των ε, επτά ετών συμφωνιών πατρική σχέση με τα κρατημέλη. Σήμερα το πρωί μίλησα για Μπράγκα, όπου μεταβήκαμε στην Πορτογαλία. Και βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με, σε μια πιο οριζόντια πολιτική. Και κάθε μέρα βγάζαμε φωτογραφίες, φωτογραφίες από επενδύσεων, Ουσιαστικά όμως όλα αυτά ε, μπαίναν, αν θέλετε, στο γενικότερο πλαίσιο όπου και να βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή που μας επαναφέρει στην ε, πραγματικότητα και όπως είπε και η κυρία Μάλετιτς, χαίρομαι που υποστηρίζουμε και την ε, πολιτική, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αισθάνομαι όπως με τα ρούχα του αυτοκρατορά. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, κάποιο άλλο σχόλιο από πλευρά των συναδέλφων, όχι. Να πω δύο λόγια από πλευρά τη Επιτροπή, ε, των μελών τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη που υποστηρίζουν αυτό το νέο εργαλείο ως μια νέα ευκαιρία. Ω τώρα λοιπόν, ναι, έχω την αίσθηση ότι το εργαλείο αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε πραγματικά. Είναι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο. χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ανάδειξει το πλήρε δυναμικό του και να αποτελέσει μια πραγματική επιτυχία, όπω αναφέρεται στον τίτλο. Δεν αφορά μόνο τα προβλήματα. Το θέμα είναι να δούμε πώς το ΕΦΣΙ θα αποτελέσει μια πραγματική επιτυχία. Αυτό είναι η πρόκληση. Η Βουλγαρία αναφέρθηκε ως μία από τις χώρες που είναι στην κορυφή των ε, επιτυχιών του ΕΦΣΙ. Αλλά αυτό οφείλεται μόνο στο χαμηλό μας ΑΕΠ. Γιατί το ΕΦΣΙ στην Βουλγαρία ουσιαστικά λειτουργεί μόνο σε ό,τι αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, λόγω της ε, τράπεζας πρόθεσης. Πρόκειται, θεωρώ, για μία από τις χαμένες ευκαιρίες της Βουλγαρίας. Μία ευκαιρία που έχει χάσει η Βουλγαρία και κάποια άλλα κρατημέλη. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του ΕΦΣΥ ήταν για κάποια από τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής ισορροπίας αυτής, αλλά και λόγω της ετοιμότητας, της προθυμίας των κρατών μελών να αποδεχτούν ένα νέο μοντέλο, να δημιουργήσουν μια εθνική πλατφόρμα και να εισαγάγουν την ευκαιρία. Συμπερίληψη επιπλέον πόρων για επενδύσεις στα κρατημέλη. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για την έκθεση αυτή, γιατί αναφέρει και περιγράφει πόσο παραπάνω δουλειά χρειάζεται για να καταστεί πραγματικά επιτυχές ε, το εργαλείο αυτό και πιο δημοφιλές. και να προετοιμάσουμε και τα κράτη-μέλη να το χρησιμοποιήσουν και να το αξιοποιήσουν μέσα στον τρόπο προκειμένου να σημειώσουν επιτυχία. Αυτό ήταν το προσωπικό μου σχόλιο ω εκπρόσωπο τη Βουλγαρία και μέλο τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Και τώρα θα σα δώσω το λόγο, κύριε Μπρικ, για να απαντήσετε στα σχόλια που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Δεν έχω σκοπό να σας πάω κόντρα. γιατί θέλω να διατηρηθεί και το θετικό και επικοδομητικό κλίμα που είχαμε κατά τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως σε τρία σημεία πέρα από αυτά που ήδη ανέφερα. Συχνά ακούμε ότι το ΕΦΣΙ 1 θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει καλύτερα, αλλά έκτοτε ε, είχαμε και το FC2, τώρα θα έχουμε το InvestEU. Το FC2, όταν ξεκίνησε και έχω μπροστά μου τα, ε, τις ερωτήσεις, τις συχνές ερωτήσεις ε, από το Σεπτέμβριο του 2017 είχε ως σκοπό να λύσει κάποια ζητήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στο FC1. Υπήρξε όμως πραγματικό benchmarking, πραγματικά ορόσημα. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε κατά πόσον αυτοί οι στόχοι που είχαμε θέσει τότε πραγματοποιήθηκαν. Και προφανώς Τώρα μόνο ε, ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και προφανώς θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όταν θα δεθεί σε εφαρμογή και το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκθεση μας έχει επίκαιρο χαρακτήρα. Και ύστερα, δύο-τρει ομιλητέ έθεσαν κάποια άλλα θέματα και η κυρία Πρόεδρος το έθεσε αυτό το θέμα ως εκπρόσωπος της Βουλγαρίας. Να εξηγήσω γιατί ακολουθήσαμε την προσέγγιση που ακολουθήσαμε για το θέμα της ε, γεωγραφικής διαφοροποίησης. Ξέρω ότι στην έκθεση μας αυτό, πριν από την έκθεση μας αυτό, το θέμα ε, απορρίφθηκε ως άσχετο, αλλά για να μην ξεκινήσουμε μια αντιπαράθεση άκαρπη, θα ήθελα να σας αναφέρω τι αναφέρεται στα καταληκτικά σχόλια και όπως είπε και ο εκπρόσωπος της ERD, η, τα συμπεράσματα αυτά του ERD τα συμφώνησαν και οι δύο πλευρές επίσης. Στα καταληκτικά λοιπόν συμπεράσματα αναφέρεται ότι όχι μόνο αποδεχόμαστε τη σύστασή μας για τη γεωγραφική κατανομή, αλλά και ότι δεσμεύονται τα κρατημέλη για κάτι ακόμα πιο ε, ουσιαστικό. Και παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕΠ θα πρέπει μέσα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΣΥ να εκτιμήσουν τα βαθύτερα αίτια των παρατηρούμενων γεωγραφικών συστημάτων και να προβλέψουν δράσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν στην υπόλοιπη ε, περίοδο εφαρμογής και θα πρέπει να εκτιμηθούν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και να εφαρμοστούν μέχρι τα τέλη του έτους 2019. Για το θέμα της γεωγραφικής διαφοροποίησης και κατά πόσον οι μέτρησεις ήταν σωστές ή όχι. Οι μετρήσει δεν θεωρούμε ότι δείχνουν την πλήρη εικόνα. Γιατί φυσικά υπάρχει η αίσθηση ότι όλα αυτά εξαρτώνται από το μέγεθος της οικονομίας. Αυτό δεν ελευθεύει όμως ακριβώς Υπάρχουν ανάγκες για στρατηγικά προγράμματα και για έργα υποδομής σε νέες περιοχές. Και όντως τα μεγάλα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα στα πλαίσια του ΕΦΣΙ. Ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια για την έλλειψη των τέτοιων προγραμμάτων στα 13 κράτη-μέλη όπου υπάρχει αυτή η έλλειψη ε, πρέπει να εξεταστούν. Σε κάποια κράτη-μέλη υπήρχαν μόνο ένα-δύο προγράμματα από το ΕΦΣΙ, από το παράθυρο για την καινοτομία και για τις υποδομές στην περίοδο μέχρι το 2018. Κάποιοι διερωτούνται γιατί να υπάρχει ανάγκη για γεωγραφική τέτοια κατανομή στα πλαίσια του ΕΦΣΙ. Καταρχάς, ε, όντως, το ΕΦΣΙ όντως αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο κινείται και βασίζεται στις ανάγκες της αγοράς. Εδώ υπάρχει μεγάλη ζητήση λοιπόν στις μεγάλα κρατημέλη γιατί είναι οι πιο μεγάλες οικονομικές αγορές. Οι εθνικές τράπεζες προώθησης είναι ουσιαστικά ενδιάμεση, συγχρηματοδοτούν και έχουν ε, προφανώς μεγαλύτερες ε, ικανότητες χρηματοδότησης σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία. Αυτό καταδεικνύει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα και των άλλων εθνικών τραπεζών πρόθεσης. Να αναφέρω επίσης και κάτι άλλο το οποίο το έζησα πρόσβατα όταν ήμουν σε μία συνέντευξη με έναν ραδιοφωνικό σταθμό της Εστονίας, οι οποίοι ε, ο σταθμός δεν μπορούσε να κατανοήσει καν ε, κατά πόσο να πήγαν καλά, πιο καλά από ό,τι αναμενόταν ή χειρότερα από ό,τι αναμενόταν. Πραγματικά δεν το κατανοούσαν. Η άποψή μας φαίνεται ότι δεν ε, συνάδει με αυτή την εντύπωση που τους είχε δοθεί. Και στη συνέντευξη λοιπόν αυτό που ανέκυψε ήταν το εξή. Κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία, κυρίω τα αριθμητικά στοιχεία στην σελίδα 37 τη έκθεση μα, βλέπουμε ότι η Εστονία είναι ένα από τα κράτη-μέλη που έλαβε τα πιο χαμηλά ποσοστά χρηματοδότηση σε απόλυτου όρου. Αυτά τα ποσά από την άλλη είναι αρκετά υψηλά είναι υψηλά σε σχέση με το ΑΕΠ τη Εστονία, προφανώς από την άλλη. Ε, κατά κεφαλήν η Εστονία είναι η δεύτερη στην ταξινόμηση με λιγότερο από 60 ευρώ άμα ε, κατά κεφαλή χρηματοδότηση, ενώ στην κορυφή είμαστε στα 120 ε, ευρώ κατά κεφαλή χρηματοδότηση. Αντί να κατηγορούμε τον έναν τον άλλον, νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε τα θέματα αυτά, αντί να εξαπολύουμε κατηγορίες. Έχουν λοιπόν δεσμευθεί πλέον για ένα μηχανισμό για να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν τις βαθύτερες αιτίε ε, τη γεωγραφική αυτή κατανομή. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο benchmarking, συγκεκριμένα ορόσημα. Δεν υπάρχει περιθώριο σε αυτό. Και υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΥ που θα πρέπει να αξιολογεί τα μέτρα που ελήφθησαν και να θέσει και η ημερομηνία υλοποίηση σε τέλη του 2019. Αυτό θεωρώ θα πρέπει να μας δίνουν ε, μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και να πω ότι όταν ξεκινήσαμε την έκθεση αυτή δεν ξεκινήσαμε να την καταρτήσουμε για να ενοχλήσουμε τον οποιοδήποτε. Αν δεν πιστεύαμε στο ΕΦΣΙ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΕΦΣΙ θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Το μόνο που μας ανησυχούσε είναι ότι το ΕΦΣΙ ενδεχομένω και να το έχει φουσκώσει λίγο ο τύπο και τα μέσα ενημέρωση. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, ενδεχομένω να έχει μεγαλύτερη εξοπιστή και μεγαλύτερο κύρο το πρόγραμμα. Τώρα, φυσικά, δεν ε, μα ενδιαφέρει τι έχει γίνει στο παρελθόν, κοιτάμε προ το μέλλον. Ελπίζουμε με την άσκηση αυτή να συνεχίσουμε την επικοδομητική εργασία στα πλαίσια του ΕΦΣΙ, προκειμένου να προσθεθεί αξία, προκειμένου να βελτιωθεί στο βαθμό που μας επιτρέπεται η χρηματοδότηση η οποία ήδη υφίσταται. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very Ευχαριστώ πολύ για την εντυπωσιακή σας πραγματικά παρουσίαση. Continue In the, in the same direction your work. Ελπίζω να συνεχίσετε τις εργασίες σας προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Και τώρα έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. And this is, uh, the exchange... Και αυτή είναι η ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Μάρκ Λεμέτρ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενικό Διευθυντή για την ε, ε ε, περιφερειακή πολιτική αλλά θα είναι εδώ σε, και δικαστική πολιτική, αλλά θα είναι εδώ σε 20 λεπτά. Σκοπεύαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην προηγούμενη ε, συζήτηση. Μπορούμε να διακόψουμε τώρα τη συνεδρίαση για 20 λεπτά ή να γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών με δύο συντονιστές. I don't think so. Maybe can I, can I ask the policy advisors to uh, check θα μπορούσα να ζητήσω από τους συμβούλους ε, πολιτικής να ελέγξουν αν μπορούν να έρθουν οι συντονιστές. Yes, please. Five, five minutes break. Πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά συντονιστές για να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ.